Ευρώπης, αλλά σίγουρα ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε πολύ, καλύτερη, πολύ καλύτερο μέτωπο απέναντι και στις χώρες αυτές. Ευχαριστώ. Ε, έληξε η συζήτηση εδώ ε, και τώρα ερχόμαστε στο επόμενο σημείο που είναι εντελώς διαφορετικού περιεχομένου. Είναι η έκθεση του κυρίου Οντή ε, αναφορικά με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δράσεις έρευνας τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης. Θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τον εισηγητή. Vous avez la parole, monsieur le rapporteur, pour 4 minutes, s'il vous plaît. Έχετε τον λόγο, κύριε εισηγητή, για τέσσερα λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, προτείνω να αφήσουμε λίγο χρόνο για να καθίσει η κυρία Επίτροπος. Σας ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, Κιούκαν Κουίν και αγαπητοί συνάδελφοι. Ο στόχος μας είναι να προβούμε σε μια αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο 2007-2013 για την έρευνα. 50 δισεκατομμύρια ευρώ το πιο σημαντικό τέτοιο πρόγραμμα στον κόσμο και άμα το συγκρίνουμε τα 17 εκατομμύρια του 2000-2006 που βέβαια ήταν πενταετές είναι πάλι σημαντική η αύξηση. Το πρόγραμμα αυτό, όπω σα είπα, ήταν 7 ετε 2007 2007-2013 και μέσα στη διαπραγμάτευση του 7ου προγράμματος πλαίσιο είχαμε τρία νέα στοιχεία που μα πρέπει να λάβουμε υπόψη στην αξιολόγησή του. Πρώτα απ' όλα βγαίνουμε από την αποτυχία τη στρατηγική τη Λισαβόνα που θεσπίστηκε από το Συμβούλιο το 2000 και ήθελε το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι η πιο ισχυρή οικονομία στη γνώση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα έχουμε τη στρατηγική 2020. Δεύτερο στοιχείο, η αποτυχία της συνταγματικής συνθήκης και τώρα έχουμε τη συνθήκη της Αβώνας με νέες αρμοδιότητες και τρίτο σημαντικό στοιχείο η χρηματοοικονομική κρίση που μας ήρθε από τις ΗΠΑ το 2008 τα νέα αυτά στοιχεία μας οδηγούν σε προβληματισμό για τα έτη 2011-2013 πρέπει να είναι τα έτη εξόδου από την κρίση αλλά μια έξοδος η οποία είναι εύθραυστη και ξέρουμε ότι οι δημόσιοι προπολογισμοί πρέπει να υπομισθούν σημαντικά κονδύλια. Είχαμε 6 δισεκατομμύρια για τα πρώτα χρόνια και μας μένουν 28,5 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να προγραμματιστούν μέχρι το 2013. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσαρμογή της πολιτικής έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα διακυβευόμενα σήμερα. Οι συνάδελφοι θα λάβουν το λόγο θα τα αναπτύξουν αυτά περισσότερο. Εγώ θέλω να σταθώ μονάχα σε δύο σημεία. Καταρχήν, απλοποίηση και αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων. Για την απλοποίηση η κυρία Καρβάλιου θα σας δώσει περισσότερα στοιχεία, χάρη στη θαυμασία έκθεσή της. Και κύριε Πίτροπε, εμεί χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την απόφαση Κομισιόν 24 Ιανουαρίου του 2011 για ένα σύστημα ενιαίας καταγραφής για τους ερευνητές θα πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο. Θα πρέπει να ξεχάσουμε τα προβλήματα του παρελθόντος. Εσείς τα γνωρίζετε πολύ καλά ως παλιό μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Έχουμε την τριετή ε, αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού που μας δίνει δυνατότητα να θέσουμε τις βάσεις μιας απλοποίησης σε επίπεδο κανονιστικό αλλά είναι αναρωτιέμαι αν το λεγόμενο <clears throat> ανεκτό ποσοστό σφάλματος είναι μια σωστή προσέγγιση. Αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ελεγκτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελεγχομένων φορών θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα μιας ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης και μιας διαδικασίας διαμεσολάβησης ώστε να μην έρχονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όλε οι διενέξει μεταξύ των ελεγχομένων φορέων και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα πρέπει, κυρία Επίτροπε, να ξεπεράσουμε αυτό το σκοπό. Έχουμε τώρα τι μεγάλε προκλήσει. Θα πρέπει να αυξήσουμε τη συμμετοχή των βιομηχανικών ομίλων μέσα στα πλαίσια της ε, πολιτικής του, της Ευρώπης του 2020 τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επίσης να τις κινητοποιήσουμε περισσότερο και για τις υποδομές θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συγχρηματοδότηση με το πρόγραμμα πλαίσιο αλλά και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πρέπει να το κάνει αυτό. Πρέπει να δώσουμε μία προτεραιότητα στην αριστεία αλλά κυρίως να βελτιώσουμε την συνεργασία των ε, υποδομών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Δεν ξέρουμε πού θα προελθούν τέτοια βραβεία Νόμπελ σε πέντε χρόνια. Τέλος για το μέλλον. Προτείνουμε στην εκθέση αυτή να διπλασιαστούν τα ερευνητικά κονδύλια για να δημιουργηθεί ο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνα που να βασίζεται σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνα. Αυτό είναι το κλειδί τη ανάπτυξη. Είναι απαραίτητο για να προχωρήσουν και οι κοινωνικέ μα φιλοδοξίε και να σεβαστούμε τι δεσμεύσει μα για το περιβάλλον. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγητά. Η Επίτροπο, η κυρία Γκόκεγαν Κίν, έχει το λόγο εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία της δήλωσης πριν την τελική ψηφοφορία αύριο. Η εφαρμογή του 7ου προγράμματος πλαισίου για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία έχει, έχει σημειώσει ορισμένα πολύ σημαντικά βήματα και προόδους. Μετά από σκληρή εργασία της ε, εισηγητρίας των σκιωδών και των υπολείπων μελών της Επιτροπής Ήτρε καθώς και της Επιτροπής Προλογισμών. Η αποτίμηση βέβαια δεν έχει καμιά σημασία αν δεν παρουσιαστούν και συζητηθούν τα αποτελέσματα ακόμη και αν δεν απορριφθούν από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους που υποτίθεται ότι εξυπηρετούν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βέβαια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο εδώ όχι μόνο γιατί μεταφέρει εμπειρίες αλλά και γιατί αναφέρει πληροφορίες από τις γνώσεις των διαφόρων βουλευτών. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Πρώτον, πρόκειται για έκθεση συνοπτική και περιεκτική που συζητά με πολύ επικοδομητικό τρόπο την αξιολόγησή μας. Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι δημιουργήσε η αξιολόγηση αυτή ανταπόκριση από όλα τα θεσμικά όργανα, ανταπόκριση η οποία τονίζει τις διάφορες πτυχές του θέματος και τις αποτιμήσεις των ανεξαρτήτων οργανισμών. Χαιρόμαστε γιατί βλέπουμε ότι αναγνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την αξία της αποτίμησής μας πολλά από τα σημεία της έκθεσης ταυτίζονται με την απάντηση της Κομισιόν για την ίδια της την αξιολόγηση. Μπορεί να μην συμφωνούμε φόλων των σημείων, αλλά το σημαντικό είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει μία βασική γενική ταύτιση απόψεων, ιδιαίτερα η αναγνώριση της ανάγκης για μια συνοπτική στρατηγική για την έρευνα και καινοτομία στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020, η ανάγκη να γίνει το πρόγραμμα πιο προσβάσιμο, πιο βατό και η ανάγκη να υπάρξουν πιο απλοποιημένες διαδικασίες ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να βασιστούν στην ποιότητα και όχι στην γραφειοκρατία. Συμφωνούμε ότι πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για την εφαρμογή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού των προτάσεων που έ, και συστάσεων που έκαναν οι αποτιμητές. Όπως είπε και η κυρία Όντι, ήδη εφαρμόσαμε τρία συγκεκριμένα προγράμματα απλοποίησης για το πρόγραμμα πλαίσιο 7, όπως την Επιτροπή Εκαθάρισης και άλλα. Ταυτόχρονα οι συστάσεις και οι απόψεις που εκφράστηκαν σε αυτή την ενδιάμεση αποτίμηση είναι ιδιαίτερα σημαντικά και για την προετοιμασία των μελλοντικών δραστηριοτήτων μας στον τομέα αυτών της ε, καινοτομίας και της έρευνας όπου απαιτείται η απλοποίηση να βασίζεται στο κοινό πρόγραμμα πλαίσιο στους νέους κανόνες και με τη βοήθειά σας στην εφαρμογή ενός κανονισμού πιο φιλικού προς τον χρήστη. Προσβλέπουμε στις μελλοντικές μας συζητήσεις και συνεννοήσεις και τα ερωτήματα που θέσατε σήμερα θα μας βοηθήσουν ιδιαίτερα. Ευχαριστώ. το της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ο κύριος Χάγλον για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Επίτροπο για τη δέσμευσή της για τα θέματα αυτά και φυσικά θέλω να ευχαριστήσω και τον εισηγητή τον κύριο Όντι. Εγώ θα παρακολουθήσω τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Προπολογισμού για τα θέματα αυτά. Θέλω να κάνω καταρχήν και ορισμένα σχόλια εξ ονόματος τη Επιτροπή Προπολογισμού. Πρέπει να πω καταρχήν ότι δυστυχώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη δική μας πλευρά ως Επιτροπής Προϋπολογισμών να βοηθηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί περικλείουν ένα τεράστιο δυναμικό δημιουργίας και ενοτομίας. Πρέπει να αναλάβουμε και ορισμένους κινδύνους για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε θετικά αποτελέσματα. Είναι, είναι απαραίτητο, κυρία Επίτροπε, να μειωθεί η γραφειοκρατία η οποία υπάρχει και πρέπει επίσης αυτή η στρατηγική να εφαρμοστεί πλήρως. Πολύ κύριε συνάδελφε. Τώρα ερχόμαστε στους ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η κυρία Καρβάλιο θα πάρει το λόγο για δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμασία έκθεσή του και για τον περιεκτικό τρόπο με τον οποίο έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό. Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη έχει μεγάλη σημασία για την ανταγωνιστικότητα και για την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού χώρου. Η χρηματοδότησή του ακόμα κατά 50% δεν έχει εκταμιευθεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι κατά το δεύτερο τμήμα, κατά το δεύτερο μέρος της χρονικής περίοδου να υπάρξει η σωστή χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Θέλω να υπογραμμίσω εδώ πέρα την ανάγκη να υπάρξει απλοποίηση της πρόσβασης στα κονδύλια, μια τροποποίηση των θεματικών προτεραιοτήτων και η προσαρμογή των κανόνων συμμετοχής για να αντιμετωπίσουμε τις νέες προκλήσεις. Η απλοποίηση της χρησιμοποίησης των κονδυλίων αυτών από τους ερευνητέ θα επιτρέψει να έχουμε σαφέστερους και διάφανους κανόνες για την απόδοση των κονδυλίων. Επομένως, στις περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να υπάρξει τροποποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού, οι απλοποιήσεις αυτές μπορούν να επιφερθούν ήδη και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για αυτά τα μέτρα τα οποία έχει ήδη λάβει προ την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, θέλω να υπογραμμίσω την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στου κέριου θεματικού τομεί που έχουν να κάνουν με το μέλλον τη Ευρώπη, όπω είναι η ασφάλεια εφοδιασμού σε ενέργεια, η υγεία και το περιβάλλον. Τρίτον, είναι απαραίτητο να υπάρξει προσαρμογή των κανόνων συμμετοχή στι νέε προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη, να έχουμε μια μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νέων ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι με τις κατευθύνσεις που έχουν τονιστεί για το επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο υπάρχει η θέληση να υπάρξει αύξηση του προϋπολογισμού στην έρευνα και την ανάπτυξη στο επόμενο οικονομικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο έτσι θα κάνουμε πιο ανταγωνιστική και πιο ευμαρή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, τώρα για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, κυρία Τόμψεν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. πολύ Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τον κύριο Ντί για την εξαίρετη συνεργασία του όσον αφορά την αξιολόγηση του 7ου πλαισίου. Ε, αντιμετωπίζουμε μία τρομερή πρόκληση απέναντι στην Κίνα, στην Βραζιλία, όπου υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Ε, θα πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι και αποτελεσματικότεροι στη δημιουργία οικονομικής ευμάρειας και ανάπτυξης μέσω της γνώσης. Αλλά αντί να ηγούμε θα είμαστε ουραγοί. Τρεις προτεραιότητες πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξουν. Πρώτα απ' όλα, απλούστευση και ξανά απλούστευση. Πρέπει να απλούστευτούν οι διαδικασίες ε, θα πρέπει να απαλληφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δεύτερο στοιχείο, ελευθερία και ευελιξία των ερευνητών. Ελευθερία να επιλέξουν το ερευνητικό κέντρο αλλά και ευελιξία με τρόπο ώστε να μπορούμε να δούμε ε, το μέλλον ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερη και αποτελεσματικότερη προσέγγιση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τόμψεν. Για την ομάδα των φιλελευθέρων κυρία Ρίς για δύο λεπτά παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Το 7ο πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης είναι το πιο σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα στον κόσμο, 54 δισεκατομμύρια για το χρονικό διάστημα 2007-2013, περίπου 9.000 ε, σχέδια χρηματοδοτούνται. Το ερώτημα είναι κατά πόσο πράγματι έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο βρίσκεται στο ύψος των επενδύσεων. Είδαμε τις προηγούμενες παρεμβάσεις και νομίζω ότι μπορεί κανείς να θέσει αυτό το ερώτημα του αν η Ευρώπη έκανε όλα αυτά τα οποία μπορούσε να κάνει. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κατακαιρματισμό στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης που ακολουθεί τον άξονα βορρά-νότου Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εξασφαλίσει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στην έρευνα και την ανάπτυξη και υπάρχουν και δυσκολίε για του ερευνητέ αλλά και τι μικρομεσαίε επιχειρήσει να έχουν πρόσβαση στα διάφορα προγράμματα. Ευτυχώ έχουμε ακόμα αισιοδοξία γιατί και το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν απόλυτη σύμπνοια στο θέμα αυτό και για την ανάγκη να υπάρξει ανακατεύθυνση τη έρευνα και τη ανάπτυξη για να αντιμετωπίσει τι μεγάλε οικονομικέ και κοινωνικέ προκλήσει όπως ελέγχθη προηγουμένως, κλιματική αλλαγή αλλά και ενεργειακή ασφάλεια, η κατάσταση με τα φουκουσιμική, όλα αυτά είναι παρά... απαραίτητα να τα λάβουμε υπόψη και επίσης να αντιμετωπίσουμε και το κολοβακτηρίδιο ασχερίσια κόλλη. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά λοιπόν, όπως τόνισε και ο κύριος Οντί, υπάρχουν οι απαραίτητες προτεραιότητες στην έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό αναφέρεται στο σημείο 9 της έκθεσής του, η Ευρώπη θα πρέπει να δώσει τον εαυτό τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει τους μεγάλους ερευνητικούς στόχους. Αναφέρθηκε ακόμα ο ότι παραμένουν 28 δισεκατομμύρια για τα τρία χρόνια που παραμένουν τα οποία θα πρέπει να κατανεμηθούν και εφόσον μιλάμε για συγκεκριμένου τομεί και για προτεραιότητε, θέλω να τονίσω την ανάγκη να έχουμε καλύτερε επενδύσει στην νάνοτεχνολογία στην η ιατρική, στα αγροτροφημικά, στις νέες ενέργειες, στην ηλεκτρονική. Μπορούμε λοιπόν φυσικά να προχωρήσουμε με τη βοήθεια των εμπειρογνωμόνων μας, αλλά η Ευρώπη μπορεί να κερδίσει τον αγώνα του πάρα πολύ μικρού. Με το... Ευρωπαίων μεταρρυθμιστών συντηρητικών, η κυρία Βίκη Φόρντ για δύο λεπτά, ε, ενάμιση λεπτό, μισής Φόρντ. Η έρευνα και η καινοτομία είναι κλειδιά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη. τα ευρωπαϊκά κεφάλαια έχουν βοηθήσει πάρα πολύ ε, και σε διακρατικά προγράμματα αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο όμω είναι το πιο γραφειοκρατικό στον κόσμο. Είναι εμφημισμένο, περιβόητο γι' αυτό. Και επίτροπε, νομίζω ότι πραγματικά μπορείτε να ε, κάνετε κάτι παραπάνω από μια απλή απλοποίηση. Ε, ο χρόνο πιέζει και θα πρέπει τα χρήματα να φτάσουν στου επιστήμονε ε, στα εργαστήρια, όχι σε αυτού που συμπληρώνουν έγγραφα απλώ. Ε, δεν μπορούν όλα να χρηματοδοτηθούν θα, και είναι δύσκολο να μετράμε κάθε φορά την προσθέμενη αξία. Αλλά δεν πιστεύω ότι ένα ευρωπαϊκό κοινό σύστημα ε, ε, αξιολόγησης της απόδοσης είναι το κατάλληλο εργαλείο. Θέλουμε επιστήμονες οι οποίοι να ανταγωνίζονται παγκοσμίω και θα πρέπει να κρίνονται και στο ίδιο επίπεδο. Η αρχή της αριστείας επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική. Το ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει κάνει περισσότερα πράγματα για την... Ε, ε, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για την υποστήριξη επιστημόνων. Αν επιλεγεί να υποστηριχθούν ομάδες επιστημόνων, δεν θα πρέπει αυτό να γίνει βάρος των, των, των επιστημόνων ατομικά. Ε, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την ε, διπλασιασμό του ευρωπαϊκού προπολογισμού σε ένα τομέα χωρίς να ξέρουμε από πού θα βγουν αυτά τα χρήματα ο προπολογισμό είναι περιορισμένο. Θα θέλαμε ε, να χρησιμοποιήσουμε με πιο ευφύ τρόπο, με κοινέ επενδύσει ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αυτά τα χρήματα. Ευχαριστώ. Τελειώσατε στην ώρα σα. Η κυρία Ματία, παρακαλώ, από την Ευρωπαϊκή Αριστερά για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω τον, τον κύριο Ντί γιατί συνεργάστηκε πάρα πολύ καλά μαζί μας ε, και το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ καλό. Η αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλησίου είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, πρέπει να επιμείνουμε στην απλοποίηση, στη διαφάνεια, στην αναδιανομή. Όλα αυτά είναι σημαντικές έννοιες στις συζητήσεις μας. Η έρευνα και η καινοτομία ε, είναι τα βασικά στοιχεία ενός πιο δίκαιου και αναδιανεμητικού αναπτυξιακού μοντέλου και πιο βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου. Αναφέρθηκαν πολύ σε κάποιες πτυχές, ε, θέλω να αναφέρω σε κάποιες πρόσθετες. Πρώτον, η αξιολόγηση απέδειξε ότι εξακολουθεί να υπάρχει υπερσυγκέντρωση των κονδυλίων σε συγκεκριμένες χώρες και σε συγκεκριμένα ερευνητικά κέντρα. Ορισμένοι κλάδοι χρηματοδοτούνται πιο εύκολα από κάποιους άλλους. Θα πρέπει να το δούμε αυτό. Θα πρέπει να εξαπλώσουμε, να διευρύνουμε τη συμμετοχή και, και στις χώρες του Νότου που αυτή τη στιγμή έχουν μικρότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι πραγματικά συμμετέχοντες ή να διευρύνουμε τη χρηματοδότηση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κοινωνία των πολιτών. Και Τέλος, ε, ε, ένα σχόλιο για το ε, θέμα της επισφάλειας της θέσης των ερευνητών. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε ερευνητές σε ορισμένα κράτη-μέλη να εργάζονται με εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εργασίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ματίας Ομπλιγκάδα. Η κυρία Τζαβέλα για ένα λεπτό παρακαλώ. Thank you, Madam σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Ντί για την θαυμάσια έκθεσή του. Το πρόγραμμα, το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και κάνουμε καλά που κάνουμε την αξιολόγηση αυτή στην, σε αυτή την ενδιάμεση φάση και χαίρομαι που ακούσα από παντού εκκλήσεις για απλούστευση των κανόνων χρηματοδοτήσεων. Δεύτερο είναι σημαντικό να ρίξουμε ιδιαίτερο φως στην ανεπαρκή συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στα προγράμματα αυτά. Ιδίω διότι η μελλοντική δημιουργία απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από αυτές. Θα υποστηρίξω επίσης τις δράσεις Μαρή Curie και θα είναι σημαντικό μέσω πρόθεσμα να αναπτύξουμε ένα μηχανισμό αξιολόγησης του μέτρου επιρροή στην αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να διατηρηθούν οι στόχοι του προγράμματος πλαισίου 7 για να επιτευχθούν εν τέλει οι στόχοι της στρατηγικής 2020. Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στους άλλους εγγεγραμμένους ομιλητές. Ο κύριος Ρόελ για δύο λεπτά παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Κυρία Επίτροπε, κύριε και κύριοι συνάδελφοι, ευχαριστώ πρώτα τον κύριο Όντι, καθώ και όλε και όλου του συναδέλφους που συνεργάστηκαν μαζί του. Η, αναθεω... ή μάλλον η επανεξέταση αυτή είναι σημαντική για τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαγάγουμε. Και θεωρώ ότι όλοι συμφωνούμε ότι η επένδυση στην έρευνα είναι κεντρική για το μέλλον τη Ευρώπη. Αν έχουμε όμω το θάρρο να συναγάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα, αυτό θα φανεί όταν θα περάσουμε στο επόμενο στάδιο. Έχουμε το θάρρος να φροντίσουμε να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδοτικά κονδύλια. Όλοι τάσσονται υπέρ, αλλά θα είναι δύσκολο. Πώς θα μπορέσουμε επίσης να δαπανηθούν τα ευιστάμενα κονδύλια με πλέον αποδοτικό τρόπο. Χαίρομαι που θέσαμε ιδιαίτερα, ρίξαμε ιδιαίτερα φως και σε σχέση με την του Καρβάγιο στην απλούστευση. Πώς θα μπορέσουμε να επιτύχουμε απλούστευση, ταχύτητα ώστε δηλαδή να αποδίδουν περισσότερο τα εφιστάμενα κονδύλια. Εκτός λοιπόν από τα επαρκή κονδύλια είναι και αυτό σημαντικό. Τρίτο, εδώ θα αντίπωσε ορισμένους συναδέλφους μου, το σύστημα ότι κατανέμω τα κονδύλια εις τρόπον ώστε ο καθένας να πάρει από λίγο δεν είναι καλό. Τα κονδύλια για την έρευνα δεν μπορούν παρά να δίδονται μονάχα με κριτήρια υπεροχής, κριτήρια αριστείας. Πώς θα διασφαλίσουμε ώστε οι χώρες εκείνες μέλη που ακόμα δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά αριστείας να μπορέσουν και αυτές ωστόσο να βασιστούν σε κάποια κονδύλια. Χρειαζόμαστε γι' αυτό άλλους μηχανισμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα μηχανισμό στο μέλλον που θα εξασφαλίσει όχι ισότιμη κατανομή των κονδυλίων, αλλά χρήση άλλων κονδυλίων στη βάση άλλων μηχανισμών. Τέλος δε, δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το ερώτημα ποια θα είναι η συγκέντρωση στα κυριότερα. Διότι αν ο καθένας ζητάει και κάτι, δεν ωφελεί αυτό την έρευνα. Πρέπει να δούμε ποια είναι εκείνα που χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη. Η κυρία Ρουέρα Μαντουρέλ για ένα λεπτό παρακαλώ. Μέχρι σε, σε ποιο βαθμό έγιναν οι αδυναμίες ε, ατού ε, με το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ε, θέλαμε να προωθήσουμε τη βασική έρευνα, αλλά και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας που στο μέλλον θα συνδυάζει τη συνοχή με την αριστεία. Ε, υποστηρίξαμε τις δράσει Μαρία Κιουρί, οι οποίε πρέπει να υποστηριχθούν περισσότερο. Αναζητούσαμε μεγαλύτερη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και με επιτυχία φτάσαμε στο 15% που θα μπορούσε να βελτιωθεί με περαιτέρω ε, απλοποίηση. Θέλαμε περισσότερη επένδυση από τον ιδιωτικό τομέα, το οποίο όμω εξακολουθεί να είναι αδυναμία, όχι μόνο εξαιτία τη κρίση, αλλά και γιατί ε, ε, ε τα τα εργαλεία που έχουμε, όπως τα CDI, ε, μπορούν να βελτιωθούν. Ελπίζω ότι με αυτή την ενδιάμεση έκθεση θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα. Ε, το λόγο ο κύριος Παναγιώτοφ θα πάρει τώρα για δύο λεπτά. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Ντί για την εργασία του είναι ένα θέμα εξαιρετικά κρίσιμο. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μπορέσει λόγω των πολλών προβλημάτων να επιτύχει τους στόχους της Λισαβόνας. Ωστόσο, στα θέματα έρευνας και καινοτομίας υπάρχουν κάποια σημεία όπου η Ευρώπη μπορεί να είναι περήφανη και που βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία. Αντιμετωπίζει ωστόσο πολλές προκλήσεις τις οποίες δεν αντιμετωπίζουν απαρατήτως οι ανταγωνιστές της και ωστόσο παραμένει ανταγωνιστική. Και αναφέρομαι στην έλλειψη φυσικών πόρων στο ευρωπαϊκό έδαφος, πράγμα που αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη της καινοτομία. Επίσης αναφέρομαι στην γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού, πράγμα το οποίο είναι ιδιαίτερο ευρωπαϊκό χαρακτηριστικό. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πιο φιλόδοξο, την πιο φιλόδοξη και δεσμευτική νομοθεσία όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Επίση, έχει ψηλά κοινωνικά πρότυπα και σέβεται τον εργαζόμενο. Νομίζω πως μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για αυτό το γεγονός, γιατί ζούμε σε μια Ήπειρο όπου ορισμένε αξίες βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού και δεν επηρεάζονται υπερβολικά από την παγκοσμιοποίηση. Κατά τη γνώμη μου, δεν μπορούμε να είμαστε η πιο βιώσιμη οικονομία στον κόσμο χωρίς σεβασμό των αξιών που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή κοινωνία. Νομίζω πως αυτό θα είναι υπέρ μας στο μέλλον. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Ζιόμπρο για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η αύξηση της καινοτομίας ε, είναι ε, βασική προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης όπως η σημερινή. Χαίρομαι που το έλαβε αυτό υπόψη του ο εισηγητής. Όμως, ε, ορισμένα θέματα ε, σχεδόν, ε, μόνο ακροθυγώς τα θίγουμε. Για παράδειγμα, δεν έχουμε αρκετές επενδύσεις στην καινοτομία στα νέα κράτη-μέλη. Πραγματικά εκπλήσει η δυσαναλογία και οι διαφορές ανάμεσα στα παλαιότερα και τα νεότερα κράτη-μέλη. Σε όλη την έκθεση αναφέρεται μόνο άπαξ αυτό το ζήτημα όμως. Δεν νομίζω ότι με αυτόν τον ε, τρόπο μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το 2007-2013 προβλέπονται παραπάνω από 80 δισεκατομμύρια ευρώ και αυτό το ποσό δεν πρόκειται να αυξηθεί. Συνεπώς θα πρέπει να αναδιανεμηθεί σωστότερα στο μέλλον. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια ε, δικαιοσύνη, λαμβάνοντα υπόψη τα νέα κράτη-μέλη, γιατί για αυτά είναι τεράστια ευκαιρία. Η επιστήμη και οι νέε τεχνολογίε θα πρέπει να υποστηρίζονται και στα νέα κράτη-μέλη, γιατί αυτό θα ωφελήσει όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το πρόβλημα της χρηματοδότησης της έρευνας είναι πιο οξύ βέβαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας ε, συνεπάγονται ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολος ο δανεισμός ε, για μακροπρόθεσμα ε, ερευνητικά προγράμματα. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Θα πρέπει επίσης βέβαια να απλοποιήσουμε διοικητικά. Η κυρία Σαρτόρη για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Οντί, καθώς και όλη την Επιτροπή της Μηχανίας για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν και για την ε, πολύ καλή συζήτηση που έγινε γύρω από αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Πιστεύω πως ε, μόνο ένα πράγμα σήμερα δεν έχει υποθεί. Δηλαδή, η αναγνώριση της συστέρησης που υπάρχει στην Ευρώπη όταν μιλάμε για έρευνα και για καινοτομία. Καλό είναι να είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματά μας, αλλά είναι ωστόσο καλό να αναγνωρίζουμε και την υστέρηση σε ορισμένους τομείς σε σχέση όχι μόνο με την παραδοσιακή, τον παραδοσιακό ανταγωνιστή μας που είναι η ΕΠΑ, αλλά και σε σχέση με πολύ δυνατούς ανταγωνιστές όπως η Κίνα και άλλες χώρες. Και πιστεύω πως η Ευρώπη αν δεν θέλει να διπλωθεί στον εαυτό της και να πεθάνει, θα πρέπει να επενδύσει περισσότερο στην έρευνα και στην ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο, μια επιλογή που δεν θα γίνει εδώ τώρα αυτή τη στιγμή. Ε, είναι μια ευρύτερη συζήτηση που αφορά τις δημοσιονομικές προοπτικές και ολόκληρο το θέμα του πώς θα χρησιμοποιηθούν οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σίγουρα είναι το πρόβλημα. Έπειτα, νομίζω πως τα θέματα που αντιμετωπίζει ο συνάδελφος Σοντή και η συνάδελφος Καρβάλιο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είναι όλα θετικά. Από την απλοποίηση μέχρι την ανάγκη συντονισμού της χρηματοδότησης, ακόμα και την απόπειρα να αναπτυχθεί η αριστεία στην καινοτομία στην Ευρώπη του 2020. Έχουμε δύο βασικούς άξονες. Ένας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπου πρέπει όντως να ευνοήσουμε την καινοτομία και εκεί την ευνοούμε με την απλοποίηση χρηματοδοτήσει και η άλλη, ο άλλος άξονας είναι τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα τα οποία δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε. Ευχαριστώ. Η κυρία Τχοτμόν, για ένα λεπτό παρακαλώ. Merci, Madame la Présidente. Madame la... Σα ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η εξαιρετική έκθεση του συναδέλφου Οντή συμπεριλαμβάνει το σύνολο των συζητήσεων με όλου του φορεί του τομέα. Δεν χρειάζεται να επανέλθω στον τρόπο με τον οποίο κρίνει ότι το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο είναι απαραίτητο αλλά πολύ περίπλοκο και γραφειοκρατικό. Θέλω να επιμείνω για δύο σημεία. Καταρχήν καινοτομία. Το, το Κοινοβούλιο έχει δεσμευτεί να προωθήσει, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να γίνει ει βάρο τη έρευνα ε, τη Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα αποτελέσματα είναι πρώτα οι και μετά είναι η δυνατότητα αξιοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων στον οικονομικό τομέα ή και στο βιομηχανικό. Πρέπει λοιπόν να γίνει σαφή διάκριση ανάμεσα στην βασική έρευνα και στην αξιοποίησή τη. Έπειτα, χρηματοδότηση. Συμφωνούμε όλοι ώστε ότι ο προπολογισμό να είναι στο ύψο των, των φιλοδοξιών που έχουμε θέσει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και συνεπεί. Δεν χρειάζεται να πολλαπλασιάζουμε τα μέσα, αλλά να τα κάνουμε πιο αποτελεσματικά. Ω προ αυτό, ο μηχανισμό ε, τη χρηματοδότηση ε, του καταμερισμού του κινδύνου είναι επιτυχή, αλλά πρέπει να είναι πιο κοντά στι μικρομεσαίε επιχειρήσει και στα ερευνητικά κέντρα. Και γι' αυτό η Κομισιόν θα πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να λύσει τα προβλήματα και να ακολουθήσει τι οδού που προτείνει η έκθεση αυτή. Κυρία Τζόρνταν Τσιζέλη, για δύο λεπτά παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο ξεκίνησε το 2007 κατόπιν της ε, διεύνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 12 νέα κράτη-μέλη. Αυτό το, αυτή η διεύρυνση δημιούργησε μεγαλύτερη διαφοροποίηση στα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι αν ε, ε, αφομοιώθηκε το πρόγραμμα από τα νέα κράτη-μέλη και αν εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής αριστείας με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, το αποτέλεσμα είναι το εξή. Μικρή συμμετοχή επιστημόνων από ορισμένα κράτη-μέλη και από ορισμένε λιγότερο αναπτυγμένε περιοχέ των, ε, των κρατών μελών. Ε, δεύτερον, ερευνητές από, μικρότερα, από τα μικρότερα κράτη-μέλη αντιπροσωπεύονται πολύ λιγότερο από την υπόλοιπη ως συντονιστές ευρωερευνητικών προγραμμάτων. Ποια είναι η εξής που μου δώσανε. Το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο βασίζεται στα κριτήρια αριστείας. Κάτι που οδηγεί στο εξοκόλουθο συμπέρασμα. Οι περιοχές οι οποίες αντιπροσωπεύονται λιγότερο σε αυτά τα προγράμματα έχουν χαμηλότερη ποιότητα ερευνητική απόδοση, απόδοση στον ερευνητικό τομέα. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να είναι αφαίρετο καλό την Κομισιόν να ε, κάνει μια ε, αξιολόγηση των παραγόντων που οδηγούν σε αυτήν την κατάσταση. Γιατί η Ευρώπη άλλωστε υστερεί το θέμα της αριστείας γιατί δεν έχουμε παρική χρηματοδότηση. Χρειαζόμαστε χρηματοδότηση και από τα διορθωτικά ταμεία Και μόνο τα κράτη-μέλη τα οποία συμμετέχουν στα διορθωτικά ταμεία θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να τα χρησιμοποιήσουν. Δεν θα πρέπει τα διορθωτικά ταμεία που ανήκουν σε ένα, τα ποσά των διορθωτικών ταμείων που ανήκουν σε μία χώρα να δίνονται σε άλλη. Η Κομισιόν σίγουρα μπορεί να λάβει υπόψη όλα αυτά. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν ελάχιστοι ερευνητέ και συντονιστέ στα προγράμματα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Ευχαριστώ από μικρέ χώρε εννοώ. Σα ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριο Κορέιαντε Ντεκάμπο για ένα λεπτό. Σα ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, θέλω να ξεκινήσω συγχαίροντας τον συνάδελφο Όντι για την εξαιρετική του έκθεση. Ακόμα και αν είναι αργοπορημένη η έκθεση αυτή, επιτρέπει να εντοπίσουμε τα προβλήματα του 7ου προγράμματος ε, πλαισίου. Η υπερβολική γραφειοκρατία, ο περίπλοκος ε, χαρακτήρας των νέων μέσων. Υπάρχει ακόμα ένας μεγάλος ε, κίνδυνος να περάσουν αυτά τα κονδύλια από το πρόγραμμα πλαίσιο σε αμφισβητήσιμα προγράμματα, πολύ μεγάλα. Υπάρχει ωστόσο και κάποιο θετικό στοιχείο, καλύτερη σχέση ανάμεσα στις διάφορες, στα διάφορα διεθνή ερευνητικά κέντρα και υπάρχουν επίσης ορισμένες περιπτώσεις επιτυχής, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μεγαλύτερη ισορροπία όσον αφορά τα φύλλα. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρξει απλοποίηση, να προωθηθεί η επιστημονική αριστεία, όχι μόνο σε ορισμένε χώρε, αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλύτερη σύνδεση του προγράμματο πλαισίου με την καινοτομία, με μέσα τα οποία θα έχουν εγκύτητα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το, όπως το πρόγραμμα ε, Eurostar το οποίο θα πρέπει να διευρυνθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ρούμπιχ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται περί της προσπάθειας ενίσχυσης της κοινότητας των ερευνητών και επομένως της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης διεθνώς. Γι' αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε ποιοι ήδη πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του προγράμματος πλασίου. Θα ζητήσω από την Ευρω... Ευρωπαία Επίτροπο να εξετάσει και το θέμα της χρήσης των προσόδων από τις ε, δημοπρατήσεις των δικαιωμάτων εκπομπών. Εδώ μιλούμε για διψήφιο αριθμό δισεκατομμυρίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευφυείς ενέργειες, για διάφορες ε, πλατφόρμες εξέλιξης μπαταριών και για άλλα προγράμματα τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν μια βιωσιμότητα του περιβάλλοντος. Αυτά μπορούν να συζητηθούν βέβαια με τον κύριο Λεβαντόφσκι καθώς και με τους αρμόδιους υπουργούς. Χρειαζόμαστε και ενίσχυση του προγράμματος CHIP όπου νομίζω το, ότι το πρόγραμμα αυτό για την τεχνολογία πληροφορικής δηλαδή έχει ανάγκη και του υλικού εξοπλισμού ώστε να μπορεί να βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Για παράδειγμα, διασυνδέσεις με οπτικές ίνες, συνδέσεις με μεσοδορυφόρων και βέβαια το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τα όσα προέκυψαν ε, μετά από τις έρευνες του 7ου προγράμματος πλαισίου να φτάσουν μέχρι αυτούς που θα τα χρησιμοποιήσουν από τους καθηγητές μέχρι τις νηπιαγωγούς. Διάδοση λοιπόν της γνώσεως από και μέσω των διδασκόντων. Το έργο είναι σημαντικό, αλλά και οι εργασίες οι οποίες επιβραβεύονται πρέπει να διατίθενται υπόψη, να τίθεται μάλλον υπόψη της ε, κοινή γνώμης. Και θα συγχαρώ και πάλι τον κύριο Ντί που δεσμεύτηκε υπέρ των μικρών και μεσών επιχειρήσεων και επίσης για τον συνάδελφο του Κάμπο που έκανε το ίδιο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Έντσου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Επίτροπε, Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Όντι για την ε, έκθεσή του, γιατί μπόρεσε να συντονίσει τις προσπάθειές μας. Πράγμα το οποίο καθορίζει και τον ε, δυνατότητά μας στην ανταγωνιστική. Πιστεύω πως ο συντονισμός και η συνεργασία στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 μπορεί να διευκολύνει και τη συμμετοχή κρατών μελών που δεν έχουν τόση μεγάλη συμμετοχή ακόμα. Συνεργασία θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να συνεργαστούν και όχι να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ε, το ποσοστό επιτυχίας που ήταν σχετικά μέτριο μέχρι στιγμή μπορεί να βελτιωθεί μέσω της απλοποίησης των διοικητικών και των δημοσιονομικών κανόνων. Επίτροπε, πιστεύω πως η γραφειοκρατία θα πρέπει να καταργηθεί. Χρειαζόμαστε απλούς και ξεκάθαρους κανόνες που θα εφαρμόζονται σαφώς. Σήμερα σας ζητώ, κύριε Επίτροπε, να μας βοηθήσετε να κινηθούμε από τα λόγια στις πράξεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Φανίστελ Ρόι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. είναι πάντα χρήσιμο να κάνει και ανείς μια ανασκόπηση του παρελθόντος, ιδιαίτερα με τέτοιου είδους εκθέσεις όπως αυτή. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την ε, ψήστης της ποιότητας δυνατή έρευνα στην Ευρώπη και θα πρέπει να την υποστηρίξουμε. Γιατί αν διαθέτουμε ευρεσιτεχνίες, οι οποίες μπορούμε να πουλήσουμε σε όλο τον κόσμο, ε, αυτό από μόνο του δεν αρκεί ε, αν τα χρήματα πάνε σε άλλα μέρη του κόσμου. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους, να έχουμε ε, πολλές ευαισθητεχνίες χρειαζόμαστε δηλαδή αριστεία, αλλά η αριστεία θα πρέπει να στηρίζεται σε δύο σκέλη, να στηρίζεται στα πόδια της και όχι να μετακινείται αριστερά-δεξιά. Θα πρέπει να έχει ρίζες σε περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πόλεις. Δεν είναι δυνατόν να εργαζόμαστε με υψηλή προσθέμενη αξία μόνο στις πόλεις όμως. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η καινοτομία, οι καρποί της έρευνας θα φτάσουν παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι θα ε, βελτιώσουν την ανάπτυξη, θα αυξήσουν την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει όλα αυτά να υποστηριχθούν με το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τα διευθυντικά ταμεία κλπ. Και βέβαια θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να βάλουν το χέρι στην τσέπη, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικά τα κοινά προγράμματα. Τώρα, δύο ακόμα ε, σχόλια. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάποιος θα αναλάβει τους κινδύνους, ότι οι κίνδυνοι θα κατανέμονται. Ε, για παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ε, δεύτερον, ναι, λιγότερη γραφειοκρατία, ασφαλώς λιγότερη γραφειοκρατία. Ας ε, δώσουμε χώρο στους ανθρώπους να καινοτομήσουν, ας δώσουμε χώρο και ευκαιρίες στις επιχειρήσεις. Δεν θα δουλέψει μόνο ο δημόσιος τομέας, δεν είναι δυνατόν να τα πετύχουμε όλα με το δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε καινούριε ευκαιρίε για το μέλλον. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μαρτσινκέβιτς για 1,5 λεπτό. E, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ ιδιαίτερο τον εισηγητή ε, για την εργασία του και τονίζω το εξή. Χρειάζεται να απλουστεύσουμε τους κανόνες και τις διαδικασίες για όλα τα προγράμματα που στηρίζουν την καινοτομία και πρέπει να εξετάσουμε τους λόγους για την τόσο ε, μικρή αντιπροσώπευση, την χαμηλή δηλαδή συμμετοχή ε, ερευνητών από τις νέες χώρες μέλη. Εάν έχουμε κοινού χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, αυτό θα εξυπηρετήσει όλους και θα επιτρέψει να στοχεύουν τις ε, έρευνές τους στις αγορές, στις ανάγκες των αγορών δηλαδή και των κοινωνιών των χωρών τους θα πρέπει να μην λησμονήσουμε και τις μικροεπιχειρήσεις και επίσης την δημιουργία τεχνολογικών πλατφορμών και κέντρων αριστείας. Οι διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης είναι ποικίλουν πολύ σε ό,τι αφορά το επίπεδο καινοτομία που επιτυγχάνουν. Οι αποκλήσει αυτέ, τα κενά μεταξύ του πρέπει να μικρύνουν και αυτό σημαίνει σωστότερη κατανομή κονδύλιων. Μην λησμονούμε και την ανάγκη συνεργειών και στο εθνικό και στο περιφερειακό επίπεδο αλλά και στο ευρωπαϊκό. Ας φτιάξουμε λοιπόν έναν αριθμό κοινών κανόνων και δημοσιονομικών ρυθμίσεων και το σύστημα κυρίως να είναι διαφανές. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να διδαχθούμε από το 7 πρόγραμμα πλαίσιο και για το μέλλον. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Χόκμαρκ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εξαιρετική του έκθεση. Πιστεύω πως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε τα εξή. Καταρχήν θα πρέπει να είναι ευκολότερο, λιγότερη γραφειοκρατία. Και αυτό το δηλώσαμε όταν ξεκίνησε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο, κατέστη λιγότερο γραφειοκρατικό και πιστεύω πως η Γράφει ε, ότι οι ερευνητές και όσοι ασχολούνται με το πρόγραμμα αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. Και νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να εμπιστευτούμε περισσότερο πανεπιστήμια που υπάρχουν εδώ και αιώνες. Δεν θα φύγουν ε, με τα χρήματα. Δεύτερον, η αριστεία. Όλη η αξία των κοινών μας προσπαθειών ότι προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ιδιαίτερη ευρωπαϊκή αξία, μια αριστεία. Όλα τα κράτη-μέλη ε, χρηματοδοτούν τους ερευνητές τους ε, και έχουμε και, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα διευθυντικά ταμεία. Αν με αυτό το πρόγραμμα δεν στοχεύσουμε στην αριστεία, θα χάσουμε την αντιγωνιστική μας πρωτοπορία στο μέλλον. Νομίζω επίσης ότι ε, με την κινητικότητα μπορούμε να πετύχουμε μέσω αυτού του προγράμματος ε, τη δημιουργία ενός ιδιαίτερου κλίματος, ε, μιας ειδική ατμόσφαιρας για την αριστεία. Και με ευτυχής που αναφέρατε την πρόταση για το ερευνητικό δελτίο στην εξασφαλιστή μια αυθόρμητη διαδικασία για την αριστεία ανάμεσα στους ερευνητές στην Ευρώπη αυξάνοντας την κινητικότητα. Και πάλι λοιπόν να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Σας ευχαριστώ. Τώρα περνάμε στο ΚΑΤΣΔΙΑ. Έχουμε 10 ομιλητές που έχουν γραφεί. οπότε θα δώσω το λόγο σε όλους, αλλά σας παρακαλώ να σεβαστείτε το ένα λεπτό. Ξεκινώ με τον κύριο Κέλλη, παρακαλώ. Συμφωνώ μαζί σας για πολλά θέματα, αλλά σήμερα είναι σαφές, Επίτροπε, ότι η Επιτροπή και τα διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου συμφωνούν. Ο εισηγητής, λοιπόν, πρέπει να επενεθεί. Αλλά όπως είπε η Κομισιόν, και εγώ είμαι ικανοποιημένος γιατί έχει δοθεί έμφαση σε ορισμένα απλά θέματα. Το πρώτο είναι η ίδια η απλοποίηση. Η ανάγκη απλοποίηση είναι ζωτική σημασία και χάρηκα που άκουσα την Επίτροπο να λέει ότι κινούμεθα προ έναν δημοσιονομικό κανονισμό φιλικό προ το χρήστη. Πρέπει να απλοποιήσουμε και επίση να εμπιστευτούμε του ερευνητέ, να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε του καλύτερου ερευνητέ, και αν το καταφέρουμε αυτό θα έχουμε και αποτελέσματα. Και τέλο δεν καταφέραμε, μάλλον αποτύχαμε με την ε, στρατηγική της Λισαβόνα. δεν μπορεί να επαναληφθεί αυτό και είναι αλήθεια ότι ε, μέσω της έρευνας ε, της επίδειξης και της απόδοσης μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντες. Λείπει. Το λόγο έχει ο κύριος Λουάν. Ευχαριστώ. Στην σημερινή συγκυρία και εν ώψη των επιτυχίας των στόχων της, ε, του 2020 θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση για να δημιουργήσουν καινούριε υπηρεσίε, καινούργια προϊόντα. Η συγχρηματοδότηση είναι πολύ σημαντική. Η πρόσβαση στις επιχειρήσεις, στις ε, ε πληροφορίες ε, ε, και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικές. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο στο οποίο να μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να υποφεληθούν από το πρόγραμμα. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη της έρευνας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, θα πρέπει να προωθήσουμε εγχειρίδια πρακτικών και να βοηθήσουμε τις ε, πολυεπίπεδες συνεργασίες. Χωρίς σαφείς διαδικασίες και χωρίς χρήσιμα εργαλεία δεν μπορούμε να πετύχουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βόν. Yeah, uh, thank you, uh, Madam President. I too would like to thank the rapporteur Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και την Επίτροπο γιατί και οι δύο είπαν ότι η έρευνα και η καινοτομία είναι σημαντικά για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και γνωρίζω βεβαίως ότι πολλά πανεπιστήμια στην Ουαλία για παράδειγμα ωφελούνται από την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να στηρίξουμε την κατάλληλη χρηματοδότηση για την έρευνα και την ανάπτυξη μέσα στον προπολογισμό της Ένωσης μπορούμε να μιλάμε υπέρ τη σηματοδότηση εδώ και να καταψηφίζουμε στην Επιτροπή του Προπολογισμού. Επίσης, είμαστε υπέρ τη απλοποίηση, ένα κοινό σύνολο κανόνων είναι απαραίτητο. Θα πρέπει ωστόσο να υπάρχει και η ευελιξία, να μην μιλάμε πάντα για καταποκοπή ποσά. Επίση, θα πρέπει να εστιάσουμε στην απόδοση. Η απόδοση είναι σημαντική, αλλά η έρευνα και η καινοτομία σημαίνει επίσης ότι πρέπει να δεχτούμε και κάποιο κίνδυνο, κάποια ανάλυση κίνδυνο. Δεν μπορούμε αυτό να το αποφύγουμε εντελώ. Και σίγουρα υποστηρίζουμε την πρόταση να δημιουργηθούν καλύτερες σχέσεις ανάμεσα στα πανεπιστήμια και στον βιομηχανικό κόσμο, ώστε να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται περισσότερο τα αποτελέσματα της έρευνας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν είναι μάθημα επιλογής. Θα πρέπει να την εξασφαλίσουμε και γι' αυτό λόγο θα πρέπει να επενδύουμε σε έρευνα και καινοτομία. Δυστυχώς, αυτοί που πιο πολλοί εποφελούνται από τα προγράμματα, χρησιμοποιούν πολλές πηγές χρηματοδότησης. Όμως αυτές οι πηγές χρηματοδότησης έχουν διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικούς κανόνες μεταξύ τους. Αυτό δυσχεραίνει πολύ την πρόσβαση στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Και δυσκολεύει και την καθημερινή ζωή όλων αυτών των ερευνητών έρευνα και η, καινοτομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να επιτευχθούν μόνο με σύγκληση, με καταπολέμηση γραφειοκρατίας και με βελτίωση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην χρηματοδότηση. Λυπούμεθα που εξαιτία της κρίσης τα κράτη-μέλη έχουν μειώσει τον ε, προπολογισμό που αφιερώνουν στην έρευνα και την παιδεία. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη να επενδύσουν στην παιδεία. Γιατί αυτό θα εξασφαλίσει και την ποιότητα της έρευνας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον συγητή, τον κύριο Ντί, που δέχτηκε την ε, τροπολογία που είχα προτείνει και καλούμε πλέον την ε, Κομισιόν να δεχτεί περισσότερα ε, μεγαλύτερη χρηματοδότηση του προγράμματος GNSS. Παρόλα άλλων, Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Γκάλαχερ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι υποστηρίζεται από πολλές πολιτικές ομάδες η παρούσα έκθεση, διότι θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει στην πρωτοπορία της έρευνας. Αυτό είναι σημαντικό. Χωρίς έρευνα δεν μπορούμε να είμαστε οι καινοτόμοι της αύριο. Χρειαζόμαστε έρευνα για να δημιουργήσουμε απασχόληση, χρειαζόμαστε έρευνα για να διατηρήσουμε την απασχόληση και να τη δημιουργήσουμε και να τη διατηρήσουμε και να παραμείνουμε ανταγωνιστική απέναντι σε αναφιόμενες οικονομίες. Χρειαζόμαστε και τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα που εγώ θεωρώ ότι είναι η κινητήρια δύναμη της ε, ανάπτυξης. Χρειάζεται λοιπόν να καταβληθούν προσπάθειες για να προσελκυστούν, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια περισσότερες μικρές και μεσές επιχειρήσεις και πρέπει να φροντίσουμε ώστε η γραφειοκρατία να περιοριστεί στο ελάχιστο. Οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων δέχθηκαν την ε, πρωτοβουλία flagship για την καινοτομία. Αλλά δεν αρκεί η στήριξη αυτή. Χρειαζόμαστε τώρα ανάληψη δράσης. Γνωρίζουμε τώρα ότι η Επίτροπος Γκέο Κέγκαν Κουίν είναι ε, άνθρωπος της δράσης. Έχουμε μηχανισμούς στη διάθεσή μας για να βοηθήσουμε να ξεπεράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την κρίση που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Όμπερμαϊερ. Ευχαριστώ. Η αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη θα πρέπει να γίνει με κριτήρια ποια είναι τα ωφέλη και ποια είναι τα μειονεκτήματα για τους πολίτες. Τα, αυτά χρηματοδοτούνται από τα κονδύλια του 7ου προγράμματος πλαισίου και θα πρέπει να κριθούν από τους πολίτες. Για κάθε πρόγραμμα, για κάθε έργο θα πρέπει να αναρωτηθούμε μπόνο, ποιος ωφελείται. Αυτό ισχύει και για τη χρηματοδότηση ερευνών για την ε, γενετική τεχνολογία, από τις οποίες έρευνες ωφελούνται μοναχά οι μεγάλες επιχειρήσεις και όχι βεβαίως οι πολίτες καταναλωτές. Χρειαζόμαστε λοιπόν αξιολόγηση πραγματική των έργων που χρηματοδοτήθηκαν, που χρηματοδοτήθηκε η έρευνά τους από χρήματα των φορολογουμένων. Ευχαριστώ. Dodge. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή για αυτή την έκθεση. Επίση ευχαριστώ την Επίτροπο που πρόσφατα επισκέφθηκε την περιφέρειά μου στη Βόρεια Ιρλανδία όπου ξέρω πω είδε κάποια υπέροχα παραδείγματα έρευνα και καινοτομία. Η οικονομία τη Βόρεια Ιρλανδία βασίζεται στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. 97% όλων των επιχειρήσεων μπορούν να ταξινομηθούν ω μικρομεσαίες. Ωστόσο είναι μια οικονομία που μένει πίσω σε σχέση με τις περιφέρειες της, του Ηνωμένου Βασιλείου και της υπόλοιπης Ευρώπης λόγω της γραφειοκρατίας όσον αφορά απορρόφηση πόρων και ε, πολλοί ανησυχούν γιατί θέλουν να μείνει ανοιχτή η πόρτα παρά όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνας και της ε, καινοτομίας. Πιστεύουμε πως είναι με σημαντική η συμβολή μας. Μεγάλες επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και βοηθούν τις μικρές για να έχουν πρόσβαση στα προγράμματα και χρησιμοποιούν αυτή την ευκαιρία, ώστε να, χρησιμοποιούν την ευκαιρία για να ζητήσω στην Επίτροπο να μας δώσει ριζικούς, παστικούς και νέους τρόπους ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να ωφεληθούν από αυτό το πολύ πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο συνάδελφος Μόλτσερ. Δεν πρόκειται γενικά περί έρευνας, πρόκειται για ιδιαίτερο πρόγραμμα έρευνας για, ε, που μας θυμίζει βεβαίως και η καταστροφή της Φουκουσίμα. Είναι γνωστό ότι το λόμπι της ε, πυρηνική ενέργειας κατάφερε πλέον πρόσφατα να περάσει την ε, ατομική πυρηνική ενέργεια ως ε, σωτήρα της ανθρωπότητας από την επιβάρυνση του κλίματος από τα καυσαέρια. Τι θα τους κάνουμε όμως αυτούς τους αντιδραστήρες όταν είναι μεν αποδοτικοί αλλά στο πρώτο παλιροϊκό κύμα καταστρέφονται και καθιστούν αδύνατο να κατοικηθούν από άνθρωπο ολόκληρες εκτεταμένες περιφέρειες και για πάρα πολλέ δεκαετίες. Η Φουκουσίμα θα πρέπει να, να σημάνει για μας μια ευκαιρία για αλλαγή νοοτροπίας. Τώρα μάλιστα που πρόκειται να συζητηθεί η ανανέωση της συνθήκης Ευρατών. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση ο κύριος Βαλέσα. Ευχαριστώ. Ακούω τα σχόλια αυτά των συναδέλφων και θα ήθελα να σας ε, μιλήσω για το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, διότι έχουμε την πράσινη βίβλο η οποία κάνει λόγο για ε, δεν κάνει λόγο για άλλους τομείς, όπως για παράδειγμα η έρευνα στο τομέα της αλίας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Ενώ ένα πλαίσιο με πολύ λίγους πόρους, μετά έγιναν και περικοπές, με αποτέλεσμα να εξαφανιστεί τελείως από το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο η αλληλευτική έρευνα. Λοιπόν, στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο, στο λάβουμε υπόψη για να αλλάξουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια και για την έρευνα στην αλία όπως προβλέπεται και από την κοινή αλληλευτική πολιτική. Η κοινή αλληλευτική πολιτική είναι πολύ σημαντική και το ίδιο και η έρευνα στον τομέα αυτό. Συνεπώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επαρκή κονδύλια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η Επίτροπος Γεωγκέχαν Κουίν. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλες και όλους ε, που συμμετείχατε. Βοηθάτε πάρα πολύ. Ε, θέλουμε να εξασφαλίσουμε ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία σε αυτό το πρόγραμμα. Στο τέλος, μέχρι το τέλος του χρόνου, πιο συγκεκριμένα 30 Νοεμβρίου, θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας ε, για τη μελλοντική χρηματοδότηση έρευνα έρευνας και καινοτομία στο πλαίσιο του ε, κοινού στρατηγικού πρόγραμματος πλαισίου. Έχουμε ήδη αρκετές ιδέες για το πώς θα πετύχουμε κάτι τέτοιο και τις εκθέσαμε στην Πράσινη Βίβλο. Ε, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε κάτω από την ίδια ομπρέλα, να υποστηρίζοντας όλη την αλυσίδα καινοτομίας από τη βασική έρευνα μέχρι την εφαρμογή στην αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή απόδοση των επενδύσεών μας. Θα, ε, Ήθελα να ακούσω την, ε, τα, τα πορίσματά σας για την πράσινη βίβλο που θα, θα αργά το καλοκαίρι. Ε, θα χρησιμοποιήσουμε πολύ τους, ε, ε, τα αποτελέσματα όλων των εκθέσεων, Καβάλιο, Ματία, Οντί κλπ. Ε, στις μελλοντικέ μας προτάσεις. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι την Παρασκευή 10 Ιουνίου οργανώνουμε μια εκδήλωση για τη λήξη της διαδικασίας διαβούλευσης πράσινης βίβλου και έχουμε προσκαλέσει αρκετά μέλη από το Κοινοβούλιο μεταξύ αυτών ορισμένους και για ομιλητές. Πάνω από 1.300 απαντήσεις πήραμε στο online ε, ερωτηματολόγιο που είχαμε στο διαδίκτυο και πήραμε και πάνω από 700 έγγραφα από εθνικές κυβερνήσεις, από ευρωπαϊκές οργανώσεις, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια, από, εθνι... από περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις κλπ. Με... που μας εκφράζουν τη θέση τους. Ε, και έχουμε πάρει τέτοιου είδους απόψεις από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς θα μας, θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ όλους σας ε, για τα σχόλιά σας και για την όθηση που δώσατε στην αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Σα ευχαριστώ, Επίτροπε. Το λόγο έχει τώρα ο εισηγητή, κύριο Οντί για δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα μάλιστα να ευχαριστήσω την Προεδρία του Κοινοβουλίου γιατί επέτρεψε τη διοργάνωση αυτή τη συζήτηση, γιατί αρχικά δεν προβλέπεται και νομίζω πω ήταν πολύ χρήσιμο που όλε οι πολιτικέ ομάδε μπόρεσαν να συζητήσουν αυτό το σημαντικό θέμα. Να πω επίση στην Επίτροπο πώς ότι είμαστε ευγνώμονες και μιλώ εξ ονόματος όλων όσων σας εκτιμούν. Έχετε μάλιστα την υποστήριξη του ε, Ιρλανδικού ε, ΕΛΚ. Ξέρετε ότι σε αυτό το θέμα ε, βασιζόμαστε σε εσά για την απλοποίηση, κύριε Επίτροπε, και για το μέγα μήνυμα που σας αποστέλνουμε. Ευχαριστώ τους εισηγητές όλων των πολιτικών ομάδων, τους συναδέλφους που κατέθεσαν πολυάριθμες τροπολογίες, καθώς και τους συνεργάτες που δούλεψαν για αυτό το θέμα, ώστε να μπορέσουμε να στείλουμε ένα ιδιαίτερο μήνυμα για τους συνεργάτες του ΕΛΚ. Απλοποίηση. Σας ευχαριστούμε και το σημειώνουμε. Οι λέξεις ανταγωνιστικότητα και βιομηχανία. Εδώ υπάρχει μια προσδοκία. Πρέπει να υπάρξει σύνδεση ανάμεσα στην έρευνα και στον εμπορικό κόσμο μέσω της ευρωπαϊκής ευρεσιτεχνίας, δηλαδή έρευνα και κοινοτομία. Η έρευνα θα πρέπει να μετατραπεί σε ανάπτυξη. Επίσης ε, και ο πρόεδρος ε, Ρέλ το ε, θύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι η καλύτερη στον κόσμο και αυτό θα το πετύχουμε μέσω της αριστείας. Αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος, επαναλαμβάνω, θα είναι ο νομπελίστες των επόμενων 5 ή 10 χρόνων. Θα πρέπει λοιπόν να τονίσουμε, να στηρίξουμε την αριστεία, να έχουμε τους καλύτερους ερευνητές του κόσμου. Χρειάζεται λοιπόν η αριστεία. Και τέλος για την χρηματοδότηση έχουμε, μας προτείνεται να διπλασιάσουμε. Μα δεν θέλουμε να διπλασιάσουμε παίρνοντα από τη Γεωργία ή από τα διευθυντικά ταμεία. Όχι, θέλουμε να συντονιστούμε καλύτερα με τα κάτι μέλη. Οι αρχηγοί των κρατών μα είπαν ότι δεν θα αυξήσουμε του ε, δημόσιου φόρου. Αντίθετα, αν συντονιστούμε καλύτερα ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα εθνικά και τα περιφερειακά που ορισμένα μάλιστα προέρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία, θα έχουμε περισσότερη συνοχή και αποτελεσματικότητα. Είχα προτείνει να θυμίσω, Πρόεδρε, είναι ένα θέμα, αλλά δεν έγινε δεκτό και πρέπει να το θυμίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο έρευνας για την αμυντική βιομηχανία. Είναι και ώρα. Τα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, επί τη βάση του άρθρου 45 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να φτιάξει, να καταρτήσει ένα μέγα πρόγραμμα για το υλικό το αμυντικό. Και επίσης σε σχέση με τη διπλή τεχνολογία. Σας ευχαριστώ και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Και τώρα, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, περνάμε στην προφορία.